Καλημέρα σας. ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Αλλά η μικρή καθυστέρηση οφείλεται σε προβλήματα κυκλοφοριακά. Πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση έχουμε ένα μικρό θέμα. Θα διαπιστώσετε ότι στην ημερήσια διάταξη συμπεριλήθηκε ένα σημείο ο δημοσιονομικός κανονισμός που αφορά το γενικό προϋπολογισμό των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ιδίω και ο εισηγητής θα μας κάνει μία επεξηγηματική παρουσίαση και αυτό το βάζουμε ως επιπλέον σημείο στη σημερινή μας ε, ημερήσια διάταξη. Αν συμφωνείτε με αυτή την αλλαγή, θα περάσουμε στα επιμέρους θέματα. Μία βιώσιμη πολιτική, θέλω να σας πω, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τον απότατο βορρά, για τον αρτικό κύκλο, είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που συζητάμε το σημαντικό αυτό θέμα στην Επιτροπή μας και αυτή η ακρόαση φαντάζεστε θα έχει παιδευτικό χαρακτήρα και νομίζω ότι εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στα θέματα που συζητάει και σχολιάζει η έκθεση Γκάλερ. Έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες μαζί μας. Θα τους δώσω αμέσως το λόγο. Και θα ήθελα να τους παρακαλέσω εκ των προτέρων να σεβαστούν το χρόνο Ξέρετε πολύ καλά ότι η λακωνικότητα είναι χαρακτηριστικό των προετοιμασμένων ομιλητών. Ο κ. Βίλ είναι ο πρώτος, Willy Ostring είναι ο πρώτος ομιλητής, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Ocean Futures στο Όσλο. Θα του δώσω πάρα αυτά το λόγο και τον ευχαριστώ βεβαίως για την παρουσία του. thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτή την πολύ σημαντική ακρόαση ε, θα ήθελα να συζητήσουμε την γεωπολιτική σκοπιά. Η γεωπολιτική σκοπιά αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ ε, του γεωγραφικού χώρου και της διεθνούς πολιτικής. Και ε, φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ στενή σχέση και εδώ λέγεται ότι εφόσον κανένα κράτος δεν είναι εκτός του γεωγραφικού χώρου κανένα κράτος δεν απαλλάσσεται από τον αγώνα για τη γεωγραφία. Ο γεωγραφικός χώρος που θα παρουσιάσω εν συντομία σήμερα το πρωί είναι η περιοχή της Αρκτικής, δηλαδή στον απότατο βορρά. Ε, η Αρκτική προκαλεί το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων κρατών, ευρωπαϊκών και ασιατικών, μεγάλων και μικρών, πολικών όπως και τροπικών και το ενδιαφέρον αυτό βασίζεται σε ε, επτά ε, βιοπολιτικά στοιχεία της περιοχής. Καταρχήν, ο γεωγραφικός χώρος ο οποίος οριοθετείται από τρεις υπήρους που αναφέρεται σε πάρα πολύ σημαντικά ε, βιομηχανικά αγαθά ιδίως ε, πετρέλαιο και αέριο μειώνεται συνέχεια ο χώρος των πάγων υπάρχει στρατηγική χρήση του χώρου αυτού υπάρχει περιβαλλοντολογική ε, ευάλωτη μορφή και Επίσης ε, ε, καλύπτεται από πολλές ε, συμβάσεις για τη διαχείριση των ωκεανών. Εδώ λοιπόν πρέπει να συνδυάσουμε, με συγχωρείτε κάτι συνέβη εδώ στο κομπιούτερ μου, πρέπει να συνδυάσουμε την γεωγραφική τοποθέτηση, της διαχωριστικές γραμμές της θαλάσσης, τις ε, θαλάσσιες οδούς και τη μείωση ε, του, των πάγων στη θάλασσα. Ε, υπάρχει υπάρχουν εμπλεκόμενα συμφέροντα της Κίνας, της Ρωσίας της ε, Ιαπωνίας και της ε, Αμερικής στο χώρο αυτό και 80% της ε, παραγωγής προκαλείται πέραν του 80ου παραλίλου και βόρεια του τροπικού του καρκίνου. Πρόκειται λοιπόν για μία βιομηχανική Μεσόγειο μεταξύ των πλέον παραγωγικών περιοχών του κόσμου μεταξύ της βορειοαμερικανικής περιοχής στον Ατλαντικό και της βορείου περιοχής του Ειρηνικού όσον αφορά το διεθνές εμπόριο μεταξύ των οικονομικών δυνάμεων αποτελεί την, ε, το πιο σημαντικό ε, γεωγραφικό ε, σύντομο δρόμο. Υπάρχουν τρεις οδοί αρκτικοί οι οποίες υπό συγκεκριμένε συνθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτόν το, λόγο. Καταρχήν το Βόρειο η βορειοανατολική διέλευση, η βορειοδυτική διέλευση από το Καναδικό Αρχιπέλαγο και η διαπολική διέλευση ε, που περνά από το κεντρικό Αρκτικό ωκεανό. Για να ε, ε, εξηγήσω τις δυνατότητες αυτών των τριών διελεύσεων θα πρέπει να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η απόσταση από τη Ιωκοχάμα στην Ιαπωνία και το Αμβούργο στη Γερμανία είναι μόνο 6.600 ναυτικά μίλια μέσω του βορειοανατολικού ε, περάσματος έναντι 11.400 ναυτικών μιλίων μέσω του, ε, της διόρυγας του Σουέζ πράγμα το οποίο σημαίνει και μία μείωση κατά 42% στην ε, απόσταση του που πρέπει να καλύψει ο ναύλος Εάν λοιπόν χρησιμοποιηθεί η διέλευση μέσω του πόλου, ε, του βορείου πόλου δηλαδή, θα μειωθεί η απόσταση αυτή κατά 700 ε, ναυτικά μίλια επιπλέον. Για να συνοψίσω, ε, το μεγαλύτερο μέρος της βορείας Αμερικανικής Δυτικής Όχθης, η Ρωσική Ανατολική Όχθη, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Κορία και η Ταϊγουάν είναι κοντύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από, όσον αφορά την απόσταση ναύλου μέσω της Αρκτικής από ότι μέσω της Μεσογείου. Και αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι οικονομικά το καλοκαίρι με 10 έως 17 ημέρες μπορούν να εξοικονομηθούν σε χρόνο ναύλου μέσω των ε, αρκτικών διελεύσεων αντί για τη διόρυγα του Σουέζ ε, για να συνδέσει κανείς τους ε, δύο παγκόσμιους ωκεανούς Βεβαίως το βασικό πρόβλημα είναι ο πάγος των θαλασσών για να μπορέσει να υπάρξει ε, μεταφορά τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αλλά τώρα η ε, η θέρμανση που οφείλεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλάζει ε, ριζικά αυτή την κατάσταση και προσεγγίζει την κατάσταση ε, της της συνθήκες πάγου του Αρκτικού ωκεανού το καλοκαίρι. Δηλαδή έχει μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα τα τελευταία χρόνια ο αρκτικός κύκλος, δηλαδή ένα χώρο μεγαλύτερο από ό,τι όλοι μαζί η Νορβηγία, η Δανία και η Σουηδία και τα τελευταία 30 χρόνια το πάχος του ε, πάγου έχει μειωθεί κατά 42%. Βάσει αυτών και άλλων επιστημονικών παρατηρήσεων υπάρχουν πρότυπα τα οποία ε, προτείνουν ότι μειώνεται περαιτέρω ο πάγος των θαλασσών κατά 30% και ο όγκος του πάγου ε, θα έχει μειωθεί 15-40% μέχρι το 2050 Υπάρχουν και άλλα πρότυπα τα οποία λέγουν ότι σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει πλέον πάγο στη θάλασσα το καλοκαίρι. Ε, το λιώσιμο αυτό των πάγων επιταχύνεται και ε, υπάρχει όλο και περισσότερη μείωση και αποδυνάμωση του πάγου των, της θάλασσας πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι παράκτιες περιοχές του Αρκτικού ωκεανού όλο και περισσότερο δεν έχουν πλέον πάγο στη θάλασσα και ε, οι ε, πλώες διελεύσεως έχουν επεκταθεί από 3 σε πέντε 6 μήνες ενώ ορισμένα σημεία των διελεύσεων ιδίως στο βορειοανατολικό σημείο χρησιμοποιούνται όλο το χρόνο για την μεταφορά στρατηγικά σημαντικών πρώτων υλών σε αγορές πιο νοτίων περιοχών. Βλέπετε εδώ την μείωση των πάγων το καλοκαίρι ενώ το χειμώνα, δηλαδή το Μάρτιο υπάρχει πλήρης κάλυψη ε, και βλέπετε ε, ε, ότι τελικά ακόμη και το χειμώνα ο πάγος μειώνεται σημαντικά. Μιλώντας λοιπόν για αυτές τις διελεύσεις, η διέλευση της ε, θαλάσσης του Κάρα, η οποία ε, βρίσκεται στη Χερσόνησο της Ταϊμύρ στην πόλη προς την πόλη του Μουρμάνσκ είναι το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα ε, της διελεύσεως για όλο το χρόνο διότι από το 1978 παραμένει ανοιχτή μέσω παγωθραυστικών 12 μήνες το χρόνο και επιτρέπει τη μεταφορά νικελίου από το Νιγκάρκα στο Μουρμάνσκ. Τα τελευταία χρόνια ε, η οδός αυτή επιτρέπει επίσης μεταφορά πετρελαίου για να εξυπηρετεί την ευρωπαϊκή και αμερικανική αγορά. Για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η διέλευση σήμερα τα παγοθραυστικά δεν χρειάζονται πλέον. Έξι ε, ε, σύγχρονα παγοθραυστικά α, έχουν τη δυνατότητα ε, να ε, μάλλον πλοία με εξοπλισμό παγοθραυστικού μπορούν ε, να λειτουργήσουν ανεξάρτητα χωρίς ειδικό παγοθραυστικό ακόμη και το χειμώνα για να διατηρήσουν ανοιχτή αυτή τη διάλευση. και αυτές οι προσδοκίες μπορούν να να πολλαπλασιάσουν στο μέλλον την ε, μεταφορά των περιφερειακών πόρων προς τις πιο νότιες αγορές και γι' αυτό το δυτικό μέρος του βορειοανατολικού περάσματος θεωρείται πολύ σημαντικό λόγω της άμεσης συνδέσεως με ε, τον βόρειο θαλάσσιο διάδρομο. Ο βόρειος θαλάσσιος ο διάδρομος ε, ε, επεκτείνεται από την ε, Λευκή Θάλασσα με συνεργασίες στο Μουρμάνκ, στο Νένετς και στο περιοχή του Αρχαγγέλ προς πολλαπλούς λιμένες στην Βόρειο Θάλασσα και ο διάδρομος αυτός θεωρείται ένα διαπεριφερειακό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσης από το 2002 και εμπλέκει εταίρους σε 22 περιοχές σε 8 χώρες. Ε, συνδυάζει ε, το ε, βόρειο θαλάσσιο διάδρομο προς την βορειοανατολική διέλευση για να συνδέσει τη βορειοδυτική Ρωσία με τον Ειρηνικό. Έχει επιπλέον ένα διατλαντικό κλάδο ο οποίος ε, συνδέει την ανατολική ακτή της Βορειοαμερικής με την Αρκτική Ρωσία. Ο κλάδος αυτός ενεργοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2008 όταν το πρώτο φορτίο πετρελαίου παρεδόθη στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε από την Αρκτική Ρωσία και επειδή το κόστος μεταφοράς πετρελαίου από το Μουρμάνσκ στη Βόρειο Αμερική είναι συγκρίσιμη με αυτή της μέση της Ανατολής ε, η θαλάσσια μεταφορά σε αυτό το κλάδο θα αυξηθεί ταχαίως στο μέλλον. Η Ισλανδία έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα για να εξυπηρετήσει αυτό το κλάδο προσφέροντας ένα λιμάνι ανοιχτής θαλάσσης, δυνατότητες επισκευών, μεταφορτώσεως φορτίου από μικρότερα σε μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα και όχι μόνο για αυτό το κλάδο αλλά και το κλάδο που συνδέει τη Βόρειο Ρωσία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ένας παρεμφερής διάδρομος μεταφοράς δεν έχει ακόμη ε, δημιουργηθεί στον ειρηνικό αλλά υπάρχουν ε, ενδείξεις ότι ένας τέτοιος διάδρομος θα καταρτιστεί ε, για να αντεπεξέλθουμε της πειρατεία των νοτίων θαλασσών και της εξάρτησης των παραδόσεων που εξαρτώνται εξαρτώνται από τις διαμάχες στη Μέση Ανατολή και αυτός που θα υποκινήσει μια τέτοια κίνηση καταρχήν θα είναι η Κίνα. Πώς λοιπόν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του παρελθόντος. Θέλω λοιπόν να ανατρέξω λίγο στο ιστορικό παρελθόν. Ένα ε, πλοίο το οποίο πηγαίνει από ε, εμπορικό πλοίο το οποίο πηγαίνει από το Άμστερνταμ στη Γιοκοχάμα μέσω του βορείου θαλασσίου διαδρόμου ε, και του βορειοανατολικού περάσματος θα χρειαστεί μόνο 400 ναυτικά μίλια δύσκολων συνθήκων πάγου δηλαδή 5 έως 6% της ολόκληρης αποστάσεως ναύλου. Ε, όταν ε, περνά από ε, τα διεθνή ύδατα που δεν έχουν πάγο ε, θα περάσει δηλαδή ένα μεγάλο μέρος από διεθνή ύδατα χωρίς πάγο και 40% ε, από ύδατα όπου μπορεί να περάσει μέσω του πάγου και στο 19ο αιώνα οι ε, Γάλλοι ε, βρήκαν έναν τρόπο να συνδέσουν την από Ανατολή με την Ευρώπη και να μειώσουν την απόσταση ναύλου δραστικά μέσω του ε, διόρυγας του Σουέζ και ε, μέσω διεθνής συνεργασίας ε, και της βελτιώσεως της ναυτιλιακής τεχνολογίας θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση του 21ου αιώνα δηλαδή να αντεπεξέλθουμε του προβλήματος της μειώσεως του, πάγου των θαλασσών. Ευχαριστώ τον κύριο Όστριγ. Ο κύριος Βάλορ, Ίγκη Μούρτζονσον, και ζητώ συγγνώμη εδώ για την κακή προφορά του δύσκολου αυτού, για μένα του, τουλάχιστον ονόματος, από την Ισλανδία, από το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας του Ρέικιαβίκ και έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Μην ανησυχείτε για την προφορά του ονόματός μου. Δεν είστε και ο πρώτος που έχετε δυσκολίες. Εγώ ασχολούμαι με τις γεωπολιτικές ε, της ε, περιοχής του Αρκτικού Κύκλου και μάλιστα υπάρχει και μια σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο. Εγώ κάνω μια εκτίμηση των πόρων επί τη βάση ε, των στοιχείων του 2008 με βάση το, την απογραφή της γεωπολιτικής υπηρεσίας σε ό,τι αφορά τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου του αρκτικού κύκλου. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα κοιτάσματα και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στον αρκτικό κύκλο είναι εντυπωσιακά και φυσικά εξετάζουμε και τις προοπτικές ε, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο στον αρκτικό κύκλο, την πρόσβαση στις φυσικούς πόρους, τη βιωσιμότητα ε, και το κατά πόσο είναι προσοδοφόρα η εξόρυξη φυσικού αερίου οι δυνατότητε πώληση και πρόσβαση στι διεθνείς αγορέ. Πάντως κυρίω ασχολούμαι με τι γεωπολιτικέ και νομικέ συνέπειε των φυσικών πόρων τη ακτική ε, περιοχή και επικεντρώνουμε σε πολλού και διάφορου παράγοντε. καταρχήν ε, αντικρώμενα συμφέροντα, συγκρούσεις δικαιοδοσίας ε, μεταξύ των αρκτικών χωρών, το ρόλο των συνθηκών του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά το δίκαιο της θάλασσας, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τα όρια τέτοιων αξιώσεων εδαφικών θέματα ακτικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά κάποιες εθνικές αξιώσεις ε, κρατών, το θέμα της πολυμέρειας και την προνομιακή θέση των ε, χωρών της Αρκτικής Ζώνης, ε, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ρωσία, Νορβηγία, Δανία, μέσω της Γρυλανδίας και το, το δυναμικό γεωπολιτικής έντασης και συγκρούσεων μεταξύ των αρκτικών χωρών αλλά υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες με συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας. Το επιχείρημά μου είναι ότι παρά τα τεράστια κοιτάσματα και το τεράστιο δυναμικό τους ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, ε, το θέμα είναι πόσο θα είναι βιώσιμη η εκμετάλλευση αυτών των κοιτασμάτων στο εγγύς μέλλον. Βέβαια, δεν υπάρχει καμία ακόμη ε, πιθανότητα ε, να κάνουμε μια μετάβαση από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Περσικού κόλπου στο ε, κοιτάσματα φυσικού αερίου του Αρκτικού κύκλου ή στα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Αρκτικού κύκλου γιατί στον Αρκτικό κύκλο υπάρχουν πολλές ε, διεκδικήσεις και αξιώσεις. Βέβαια υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών ε, μια και υπάρχει όμως ε, μια κοινότητα ασφάλειας ε, μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών, πιστεύουμε ότι η διαμάχη, η διαφυσβήτηση μάλλον δεν θα πάρει τεράστιες διαστάσεις. Άλλωστε υπάρχει συμφωνία ήδη για το βόρειο δυτικό πέρασμα και με το βόρειο πέρασμα για τη Ρωσία αφορά εσωτερικά ύδατα. Αλλά υπάρχουν και, υπάρχει ένα τμήμα που είναι διεθνή ύδατα. Στην έκθεση μου επιχειρηματολογώ ότι κάποιες επικαλυπτόμενες αξιώσεις εδαφικές δεν χρήζουν άμεσες λύσεις. Κατά πάσα πιθανότητα θα καθυστερήσουν την ανάπτυξη την εκμετάλλευση των πόρων μάλλον. Παρ' όλα αυτά η αμφισημία της ε, διακυβέρνησης εξαιτία έλλειψης μηχανισμού διακανονισμού των διαφορών ε, υπάρχουν προβλήματα γιατί υπάρχει ε, κάποια βεβαιότητα σε ό,τι αφορά τα επτά αρκτικά κράτη. Αυτή η εμφυσιμία σε ό,τι αφορά την αρκτική διακυβέρνηση οφείλεται σε πολλούς και διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, η συνθήκη του ΟΗΕ για τα όρια της ε, υπηρετικής υφαλοκρηπίδας και το μέγεθός της η συνθήκη του ΟΗΕ δεν ε, προβαίνει σε διακανονισμό των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν συστάσεις, γίνονται κάποιες συστάσεις προς τα πέντε αρκτικά κράτη και σύσταση για διαπραγμάτευση προκειμένου να διαθετηθούν οι διεκδικήσεις τους. Και υπάρχει και κίνητρο ε, για τα κράτη αυτά να καταλήξουν σε φιλική λύση και διακανονισμό, αλλά δεν αποκλείεται και σύγκρουση μεταξύ τους, θεωρητικά. Ο ρόλος του Αρκτικού Συμβουλίου είναι ότι είναι απλώς συμβουλευτικό όργανο και δεν ε, λαμβάνει αποφάσεις. Έχει περιβαλλοντικό έργο, και ενισχύει την πολυμερή συνεργασία. Παρ' όλα αυτά δεν έχει αρμοδιότητα για θέματα πολιτικά ή θέματα ασφάλειας στην αρκτική περιοχή. Και έχει εξεταστεί το κατά πόσο θα θεωρείται ο βασικός φορέας για τη διαχείριση των αρκτικών θεμάτων. Αν έχει λόγο δηλαδή στα θέματα εκμετάλλευση φυσικών πόρων ή διακανονισμού διαφορών. Το, η πιο επίμαχη πρωτοβουλία ήταν η απόφαση των πέντε αρκτικών ζωνών ε, να τονίσουν τον προνομιακό τους ρόλο στην περιοχή, στην συμφωνία, στην συνεδρίαση του Λούλισαντ ε, το 2008. Πάντως, ε, η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή δεν μπορεί να γίνει με εξαίρεση της Ισλανδίας, Φιλανδίας και Σουηδίας των τριών αρκτικών ε, χωρών ή με αποθε... περιθωριοποίηση των γηγενών πληθυσμών. Η καναδική κυβέρνηση έδωσε μια συνέχεια το Μάρτιο του 2010 στην πρώτη συνεδρίαση του 2008 και συγκρότησε μια νέα συνεδρίαση των πέντε αρκτικών χωρών. Αλλά και αυτή ήταν αποτυχημένη κατά κάποιο τρόπο γιατί η Χίλαρη Κλίντο για παράδειγμα, η Αμερικανίδα υπέξ επέκρινε την ε, καναδική κυβέρνηση που δεν προσκάλεσε και τους υπόλοιπες ε, ενδιαφερόμενους, ε, τις ενδιαφερόμενες χώρες στην περιοχή. Δεν υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά αυτές τις πέντε χώρες για την αρκτική διακυβέρνηση. Και υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της ανάγκης αυξανόμενης συνεργασίας μεταξύ των αρκτικών χωρών για να αποφευθούν να αποφευθεί κλιμάκωση των εδαφικών διαμαχών. Ανακεφαλώνοντας, θα ήθελα να πω ότι σήμερα με την κατάσταση στην αρκτική ζώνη βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση για ετοιμότητα, όχι από στρατιωτική άποψη, αλλά από πολιτική και νομική. Για να γίνει με σωστή ερμηνεία αυτής της περιοχής. Δεν υπάρχουν πολλές εντάσεις στην αρκτική ζώνη. Βέβαια υπάρχουν ε, πολλοί δημόσιοι φορείς ε, και πολλές χώρες, αλλά που τηρούν το διεθνές δίκαιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επικαλυπτόμενα συμφέροντα και μερικές φορές εθνικιστικές δηλώσεις δεν εξυπηρετούν το στόχο της διαπεριφερειακής και μακροπρόθεσμης συνεργασίας. Ιδιαίτερα όταν πλησιάζουμε στη φάση της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. Θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο, φτάνοντας στο τέλος της παρέμβασής μου. Μερικές φορές, ακόμη και αν η αρκτική ζώνη είναι ζώνη χαμηλών εντάσεων, μερικές φορές κάποιες ε, δηλώσεις ε, μπορούν να δημιουργήσουν πολιτική πραγματικότητα. Όταν οι Ρώσοι έβαλαν σημαία στο βυθό του Βορείου Πόλου, δημιούργησαν ε, μία αναταραχή, γιατί μπορεί η χειρονομία τους να είχε λόγους εσωτερικής πολιτικής και κατανάλωσης, αλλά παρόλα αυτά δημιούργησαν τη δράση στον Καναδά, ή επιτάχυνε την αρκτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών που εξέδωσαν και ένα ανακοινωθέν σχετικά. Από αυτή την άποψη λοιπόν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι δηλώσεις που μπορούν να γίνουν στον τομέα αυτό ίσως διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στο μέλλον. Το ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά και η τελευταία παρουσίαση για το θέμα αυτό θα γίνει από το James Reynolds από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος του Αρκτικού Συμβουλίου. Uh, Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να παρουσιάσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την Αρκτική Ζώνη. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχει ε, ένα προσανατολισμό προς την περιοχή για τρία μέρη. Τρία μέλη της είναι, της της, ανήκουν στην Αρκτική Ζώνη και συνδέονται και με την Νορβηγία, τη Γρυλανδία κτλ. Και επομένως οι πολιτικές μας όπως η έρευνα συνδέονται με την Αρκτική Έχουμε δώσει 200 εκατομμύρια ευρώ πέρα από τις συνεισφορές των μελών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το περιβάλλον, ε, οι γηγενείς πληθυσμοί, οι μεταφορές, η ενέργεια και η θαλάσσια πολιτική. Επίσης δραστηριοποιούμαστε σε διάφορους τομείς που αφορούν την Αρκτική, κυρίως η βόρεια διάσταση Επίσης η συνεργασία για την Αρκτική και η σύμβαση ΟΣΠΑ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορείου Ατλαντικού που περιλαμβάνει και την περιοχή που περιγράφτηκε από τον καθηγητή Έστρομ. Ανήκει στην περιοχή αυτή ΟΣΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλόμενο μέρος. Πέρα λοιπόν από τους, τους οικονομικούς δεσμούς υπάρχουν και αυτοί οι θεσμικοί δεσμοί που συνδέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αρκτική Ζώνη. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά διαμορφώνει μια αρκτική πολιτική. Ταυτόχρονα αναγνωρίζει το θεμητό συμφέρον των μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ανήκουν στην Αρκτική να έχουν συμφέροντα. Το Συμβούλιο των Υπουργών στα συμπεράσματα του 2009 καθορίζουν σαφείς προτεραιότητες για να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν την Αρκτική σε συνεργασία με τους πληθυσμούς της και να υπάρξει βιώσιμη χρήση των πόρων της. Επίσης θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στην ενδυνάμωση της πολυμερούς διακυβέρνησης που θα βασίζεται στις υπάρχουσες συμβάσεις και κυρίως τις συμβάσεις, τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και να διερευνήσουμε τρόπους για να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις για τη ζώνη αυτή. Αναγνωρίζουμε το βασικό ρόλο του Αρκτικού Συμβουλίου και την ε, σημαντική δουλειά που έχει κάνει και οι ομιλητές οι προηγούμενοι ε, μίλησαν ε, για το ρόλο του που έχει στη διαμόρφωση των αποφάσεων, όχι στη λήψη των αποφάσεων και στη σημαντική επιστημονική δουλειά του. Και νομίζω ότι ακριβώς εκεί η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει